με την έκθεση του συναδέλφου Βαλκάρ Σελσίσο Καθίστε σιγά σιγά Έχουμε ονομαστική ψηφοφορία Συνάδελφος Ντάρτμοντ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω αν μπορούμε να συγχαρούμε τον πρώην Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόζο, για το διορισμό του στην Golden Sachs. Επίσης, θέλω να εκφράσω και την ανησυχία μου, διότι η σύνταξή του ως πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής δεν του αρκεί. Δεν ξέρω αν ε, είναι κατάλληλος ο χώρος για να το κάνουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε, αυτό. Πρόεδρος, για το πρώτο τμήμα της ερώτησής σας, ε, το ερώτημα, και δεύτερον, ε, για τη δεύτερη απάντησή σας υπάρχουν κανόνες σχετικά. Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Μιχαήλοβα. Άρχεται η ψηφοφορία, πάλι ε, ονομαστική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση της Άλμπα Μπίντεγκάιν και Γιάννη Κεμπράντι. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση της Βιέφκα. Ψήφι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έκθεση Χαουτάλα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έκθεση Λουμποχετό, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έκθεση Γιούλιο Βίνκλερ, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Έκθεση θα λοιπόν Μπίντεγκάιν, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Έκθεση Σόλτες. Έχουμε τρεις εκθέσεις του συναδέλφου Σόλτες. Έχετε το λόγο, συνάδελφε. Δεν βλέπω που κάθεται όμως. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πριν από την ψηφοφορία για τους υποψηφίους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα ήθελα να υπογραμμίσω τα εξής. Βλέπουμε ότι το Συμβούλιο πρέπει να, να, να εγκρίνει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν πρότασης των ε, κρατών μελών. Το, Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο παίζει λοιπόν συμβουλευτικό ρόλο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το Συμβούλιο δεν μπορεί να ελέγχει και την βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και αυτό που έχει συμβεί σε προηγούμενες περιπτώσεις και για το μέλλον, ε, πιστεύω πως το Συμβούλιο πρέπει πραγματικά σοβαρά να σέβεται τη θέση και τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν πρόκειται για αυτές τις υποψηφιότητες. Δεν ξέρω γιατί ακολουθεί τέτοια διαδικασία εφόσον στο τέλος θέλει να κάνει εκείνο ό,τι του αρέσει ε, και μόνο. Καλύτερη λοιπόν ε, διαβούλευση θα πρέπει να γίνεται. Δεύτερον, οι υποψήφοι στο ελεγκτικό συνέδριο και πάλι μόνο άνδρες. Θα πρέπει ακόμα μια φορά να, να τονίσουμε την σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στα φύλλα. Γι' αυτό και θα πρέπει να καλέσουμε το ελεγκτικό συνέδριο στο μέλλον να σέβεται την ισορροπία ανάμεσα στα δύο φύλλα. Υπάρχουν μόνο τρεις γυναίκες μέλη ε, στο σύνολο των ε, ελεγκτών. Και ο αριθμός των μελών δεν μπορεί να μειώνεται διαρκώς. Θα ελπίζω πως αυτές οι αρχές θα γίνουν σεβαστές στο μέλλον. Ευχαριστούμε τον κύριο εισηγητή. Τώρα ακολουθούν τρεις ονομαστικές ψηφοφορίες. Ξεκινάμε. Α, ζητώ συγγνώμη. Ε, μυστικές ψηφοφορίες, όχι ονομαστικές. Ξεκινάμε με τον κύριο Λάζαρο Σταύρου Λαζάρου. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα, μυστική ψηφοφορία για τον κύριο Ζωάου Φιγκερέιντο. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ακολουθεί η μυστική ψηφοφορία για τον κύριο Λεό Μπρινκάτ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα, περνάμε στην έκθεση Λάγκε. Εγκρίνεται με βάση τη Συμφωνία Συμβουλίου Κοινοβουλίου. Έκθεση Κάπελ. Ε, για το πρώτο μέρος, ψήφι υπέρ. Κατά. Λίγοι συμμετέσχουν. Άρχεται η ψηφοφορία για να το ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. να ε, ψηφίσουμε και την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Λάγγεν. Παράγραφος 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 22, πρώτη τροπολογία, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 23. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 24 σε δύο τμήματα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 30 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 44 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφο 48 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 49. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 51 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περάγραφος 53 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 54 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές,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 Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 66 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 70 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 71 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 72 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 73 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη G υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα στο σύνολό του όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Γκίχεκ, παράγραφος 9, υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. μου λείπουν οι αντιρρήσεις από την ε, ε, ομάδα ΙΑΤΕ. Παράγραφος 23. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Εψήφισαν όλοι. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 28 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 31. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 39 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 41 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 45, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 48 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 51. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορία; Εγκρίνεται. Παράγραφο 52 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφο 55 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Παράγραφος 56 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Παράγραφος 69 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Παράγραφος 92 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Παράγραφο 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη κάπα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη τάφ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη β σε δύο τμήματα. Πρώτον, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Μισό λεπτό, κυρία Φωνστόρφ. πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η κυρία Φωνστόρφ για διαδικαστικό θέμα. Ε, δοκιμάστε το, νομίζω ότι λειτουργεί. Κύριε Πρόεδρε, κάνετε μια παρατήρηση κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο σημείο του κανονισμού βασίζεστε γιατί θα έπρεπε ο ΓΟΥΙΠ από την ομάδα της, ε, των Σοσιαλδημοκρατών να συμμετέχει. Κυρία Φωνστόρ, κύριε συνάδελφε, δεν είπα ότι έχω δυσκολίες. Είπα ε, ότι ε, ήταν πιο εύκολο να παρακολουθώ τους συναδέλφους ε, κατά αυτόν τον τρόπο χωρίς το WIP. Έκθεση Νταμάτο. Άρχεται η ψηφοφορία, μονομαστική ψηφοφορία. Τα ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Μπρεσό. Παράγραφος 7. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 31. Ε, μια προφορική τροπολογία της κυρίας Μπρεσό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προφορική τροπολογία εισάγει την στήριξη για το συντονισμό των υπηρεσιών διάσωσης σε, στις ορεινές περιοχές Mount Rescue Services ε, στην περιοχή των Άλπαιων. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κανείς ε, κατά. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Να ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται με την τροπολογία. Μετά την παράγραφο 36, ονομαστική ψηφοφορία για το πρώτο, την πρώτη τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερη τροπολογία, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τρίτη τροπολογία, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 43, τέταρτη τροπολογία, με ονομαστική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 47 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος, το σύνολό του όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι, πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Κοράο, παράγραφος 2 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 4 μια προφορική τροπολογία του κυρίου Κοράου. Ich glaube, it works. No, not working. Okay. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αλλάξω την προφορική τροπολογία. Υπάρχει στο τέλος του καταλόγου ψηφοφοριών σας.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 Παράγραφος 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 11 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 12 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 13 προφορική τροπολογία του κυρίου Κοράου στο αρχικό κείμενο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και πάλι θα ήθελα να μεταφέρω την τροπολογία που θα τη βρείτε και πάλι στο τέλος του καταλόγου με τις ψηφοφορίες. Αν θέλετε μπορώ να σας τη διαβάσω. Υπάρχουν αντιρρήσεις, ρωτάει ο πρόεδρο, Δεν υπάρχουν υπέρ, κατά, απόχέ, Εγκρίνεται. Παράγραφος 14. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ. Απορρίπτεται. Παράγραφος 15. Προφορική τροπολογία. Πού και πάλι την έχετε στον κατάλογο, κύριε Κοράου. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ η προφορική τροπολογία καλύπτει την ε, ε, ψηφοφορία κατά τμήματα για τη λέξη particularly και θα βρείτε στο τέλος του καταλόγου ψηφοφορίας την προφορική τροπολογία. Μπορώ να σας τη διαβάσω αν έχετε χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Κοράουλη, ο Πρόεδρος. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία. Έχουμε... Δεν χρειάζεται σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε και το συνολικό κείμενο, λοιπόν. Μετά την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 17 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, τρίτο τμήμα, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 20 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, απόχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφος 24 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Παράγραφο 26 υπέρ. Α, να το τρίτο τμήμα της 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 32 με μια προφορική τροπολογία του κ. Κοράου. Ε, νομίζω ότι ξέρετε τι θα σας πω. Θα ήθελα να δείτε την προφορική τροπολογία στο κείμενο στο τέλος του καταλόγου ψηφοφοριών. Ευχαριστούμε κύριε Κοράου. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται.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 Το σύνολο του τροποποιηθέντος ψηφίσματος σε ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασες της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην τελευταία ψηφοφορία, συναδέλφων Σντάνοκα και Χιούτε. Παράγραφος 3 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέραση τη ψηφοφορία.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 να ελέγξουμε το τέταρτο τμήμα της 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Για το... Παράγραφος 6. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 7 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφο 8 σε 3 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10 με δύο τμήματα. Με ονομαστική ψηφοφορία το πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα Άρχεται η ψηφοφορία, με ονομαστική ψηφοφορία και πάλι. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφο 15 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Παράγραφο 18, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφο 20 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Παράγραφο 21 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Παράγραφος 23 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Παράγραφος 24 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Κυρία Φων Στόρκ, δεν ψηφίσατε υπέρ. Παράγραφος 26 υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε. Πολλές αποχές νομίζω. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 28 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, είναι για το αρχικό κείμενο. Εγκρίνεται επομένω. Τέταρτο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έκτο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έβδομο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όγδοο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές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 Παράγραφος 35 σε τέσσερα τμήματα, όλα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται για το πρώτο τμήμα η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 37 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 41 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Πολλές αποχές να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφο 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 46. Σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 47 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 49 σε τρία τμήματα. Το πρώτο με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 51. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 52. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται.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 Πέρα τη ψηφορία απορρίπτεται. Παράγραφο 55 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφος 56 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. Παράγραφο 59 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία.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 Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Δέλτα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ε σε δύο τμήματα και η δύο με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται για το πρώτο τμήμα. Εψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Ζ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Ι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται.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 κατά, αποχές, απορρίπτεται. αιτιολογική σκέψη. Θέλετε να ελέγξουμε το μη. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Ζήτω συγγνώμη. Αιτιολογική σκέψη Q σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη S σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη τάφ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Β σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ΑΒ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ΑΕΦ. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ΑΓ. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ΑΙ υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για το ΑΙ. Εψήφισαν όλοι. Πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα πριν ψηφίσουμε για το σύνολο του ψηφίσματος, θα ήθελα να σας παρακαλέσω ε, όποιος δεν θέλει να παρακολουθήσει τις αιτιολογήσει ψήφου, να βγει γρήγορα από την αίθουσα, ε, από σεβασμό για του συναδέλφους που θέλουν να ακούσουν. Άρχεται η ψηφοφορία τώρα για το σύνολο του ψηφίσματος. Σε ψήφισαν όλοι. Ε, τώρα τελείωσε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Meine Damen und Herren, wir kommen zu den Stimmerklärungen. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στι επεξηγήσει ψήφου. Ε, ξέρετε ότι ο πρόεδρο για τον συνάδελφο Κόλβιν Μίκε ε, τον έχει αποκλείσει από την ε, επεξήγηση ψήφου.